την Πρόεδρο τη Επιτροπή και είπα τη εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια για το θέμα τη Ουκρανία. κυρία Άστον όμω δεν μπόρεσε να μείνει μαζί μα σήμερα, οπότε εξ ονόματό τη θα παρουσιάσει το θέμα ο Επίτροπο Στέφαν Φούλε. Mr. Chairman, thank you very much for this. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Άστον, η οποία μου ζήτησε να σας μεταφέρω αυτά τα οποία σκόπευε να σας πει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να κάνω μια δήλωση για την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία. Θα ήθελα να κάνω τις παρατηρήσεις μου εν ώψη τριών σημαντικών γεγονότων. Έχουμε την υπουργική διάσκεψη με την Ουκρανία που θα λάβει χώρα 26 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Τις τοπικές εκλογές θα λάβουν χώρα στις 31 Οκτωβρίου και την 14η Σύνοδο κορυφή με την Ουκρανία που θα λάβει χώρε Βρυξέλλε 22 Νοεμβρίου. Πρόσφατα η Ουκρανία βεβαίω απολαμβάνει υψηλό επίπεδο πολιτικών ελευθεριών. Οι διαδοχικές εκλογές θεωρήθηκε πω έλαβαν χώρα σύμφωνα με τι διεθνεί προδιαγραφέ. Έχει αναπτύξει λοιπόν μια δυναμική κοινωνία των πολιτών και ΜΜΕ και έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως συνέπεια αυτών των εξελίξεων και της δέσμευσης διαδοχικών κυβερνήσεων για στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις με την Ουκρανία έχουν αποκτήσει σημαντική όθηση. Αυτό αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στην φιλόδοξη συμφωνία σύνδεσης ε, την οποία διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή και στόχο έχει να επιτύχει το διπλό στόχο της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση του Πρόεδρου Γιαννόκοβιτς έχει ξεκινήσει μια σειρά σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες που πρέπει να επενέσουμε. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την υιοθέτηση νομοθεσίας δημοσίων προμηθειών που θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Υιοθέτηση νομοθεσίας μεταρρύθμισης του τομέα του φυσικού αερίου, κατά το οποίο βέβαια το έδαφος για την ένταξη της Ουκρανίας στην ενεργειακή κοινότητα και βέβαια υπάρχει μια συμφωνία παροχής βοήθειας από το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο το οποίο διασφαλίζει μακροοικονομική σταθερότητα, διαφάνεια και επιστροφή στην ανάπτυξη. Αυτά πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση και πρέπει να συνεχιστούν. Η Ουκρανική κυβέρνηση επίσης κατάφερε να επιτύχει ένα επίπεδο σταθερότητα το οποίο δεν είχε επιτύχει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι μια σημαντική και απαραίτητη εξέλιξη για να διασφαλιστεί αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ανησυχούμε για τις πάρα πολλές αναφορές όσον αφορά την επιδείνωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Ουκρανία. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι αυτά τα οποία ακούγονται για την ελευθερία των ΜΜΕ την ελευθερία του συνεταιρίζεται και του συνέρχεστε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ο σεβασμό αυτών των βασικών ελευθεριών είναι ουσιαστική σημασία, είναι η καλύτερη εγγύηση των ατομικών ελευθεριών. Εξασφαλίζουν γνήσιο ανταγωνισμό των ιδεών, είναι ουσιαστικό συστατικό μέρος των καινοτόμων και ανταγωνιστικών κοινωνιών. Την 1η Οκτωβρίου το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας εξέδωσε μία απόφαση που ανέτρεψε τις συνταγματικές αλλαγές που είχαν γίνει μετά την Πορτοκαλή Επανάσταση του 2004. Η απόφαση αυτή αυξάνει την ε, ανάγκη επίτευξης ε, ευρύτερης συνταγματικής μεταρρύθμισης της Ουκρανίας μέσω μιας διαδικασίας μεταρρυθμιστικής και αντικατοπτρίζεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου τρέχοντος για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των εξουσιών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μας ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών ε, και το κράτος είναι οι βασικές αρχές που μας ενώνουν, είναι αρχές οι οποίες δεν στις οποίες δεν χωράει συμβιβασμός. Το ίδιο και για τις σχέσεις μας με εταίρους κλειδιά όπως η Ουκρανία. Ο ρυθμός προσέγγισης με την Ουκρανία θα κριθεί από τον πλήρη σεβασμό αυτών των αξιών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και τώρα περνάμε στου ομιλητέ, οι οποίοι θα μιλήσουν εκ ονόματο των διαφόρων κοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Μάικλ Γκάλερ εκ μέρου του ΕΛΤ, για πρώτος ομιλητής για δύο λεπτά. Für eine europäische Zukunft des Landes hat sich das ukrainische Volk immer wieder eindrucksvoll ausgesprochen. Ευχαριστώ. Ακούστηκαν ε, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις οι οποίε ομακρύνουν τη χώρα αυτή από την Ευρώπη, κάτι το οποίο αναμέναμε βεβαίω πριν από τις ε, δημοτικές ε, εκλογές ε, και βεβαίω έχουμε και την σύνοδο κορυφής η οποία πλησιάζει οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ελευθερία του τύπου καθώ πλησιάζουμε προς εκλογές δεν είναι δυνατόν αυτά να εξισωθούν ή να αντισταθμιστούν από τις θετικές οικονομικές εξελίξεις μιλάμε για περισσότερο κινέζικο παρά ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ε, κοινωνίας. Βεβαίως όλα αυτά δεν τα γνωρίζει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ούτε δικαιολογούνται επειδή υπήρχαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση ανάλογα προβλήματα. Δεν υπήρχε ούτως ή άλλως ε, παραδείγματος χάρη επίσκεψη των μυστικών υπηρεσιών στον πρίτανη του καθολικού ε, πανεπιστημίου της χώρας, ούτε κατά κατασχέσεις υπολογιστών, ε, δηλαδή όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε λαμβάνουν χώρα. Οι γνωστές μέθοδοι των μυστικών υπηρεσιών. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργούσουν μια αυτοκρατορία των ΜΜΕ, η οποία επίσης απομακρύνει την Ουκρανία από την Ευρώπη. Δεν έχουν απομείνει λοιπόν πάρα πολλά πράγματα να κάνει η αντιπολίτευση στις, ε, στις δημοτικές εκλογές και βλέπουμε και διάφορα άλλα κόμματα μαριονέτες που δημιουργούνται. Στο Κίεβο δε καταρχούνται εκλογικές περιφέρειες για να μην λάβουν χώρα οι εκλογές με στόχο να υπάρχει έλεγχος των περιοχών εκείνων που διαφωνούν με την κυβέρνηση. Βεβαίως τα κράτη, μας, ε, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη δημοκρατική συνένεση και στο σεβασμό της αντιπολίτευσης υπέρ του κράτους δικαίου, υπέρ της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Ε, για όλα αυτά επιθυμούμε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο η Ουκρανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλε. Ο κύριος ε, Μιχάλησκι έχει σηκώσει μια γαλάζια κάρτα, ένα γαλάζιο χαρτί. Αυτό τι αφορά, θέλετε να ερωτήσετε κάτι τον κύριο Γκάλερ. Α, ωραία. Δέχεστε να ακούσετε τώρα τον κύριο Μιγάλης και κύριε Γκάλερ. Ωραία. Παρακαλώ κύριε Μιγάλης και έχετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Μικρόφωνο. Παρακαλούμε με μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ που δεχθήκατε το ερώτημά μου. Πάντοτε είναι ευχάριστο να ε, είναι δυνατή, να, δυνατό να υπάρχει συζήτηση. Η πολύ μελανή περιγραφή της κατάστασης ε, στην Ουκρανία σήμερα, την οποία συγκρίνεται ακόμη και με την κατάσταση στην Κίνα. Ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με αυτό. Θεωρείτε ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα ώστε θα πρέπει να ε, κατηγορήσουμε με τόσο αυστηρά λόγια σήμερα την Ουκρανία. Έχετε 30 δευτερόλεπτα κύριε Γκάλερ για να απαντήσω τον κύριο Μιγκάλσκι. Αυτό που είπα ήταν ότι όσον αφορά την οικονομική ευμάρεια προσπαθούν να την πετύχουν μέσω πολύ αυταρχικών τρόπων. Δεν είναι ευρωπαϊκός τρόπος. Το ξέρουμε αυτό από την Κίνα. Δεν κάνουμε παραλληλισμό. Θα ήταν ασφαλμένη προσέγγιση λέμε. Ευρωπαϊκή προσέγγιση πάντως δεν είναι. Και η εικόνα που σκιαγράφησαν είναι πολύ ρεαλιστική για εκείνους που ζουν εκεί πέρα. Και αυτό το οποίο πρέπει να ευχθεί έχει ακόμη δρόμο. Ευχαριστώ. Τον λόγο Ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο σε ένα λεπτό. Γι' αυτό και δεν ξεκινώ τώρα συζήτηση για αυτό το θέμα. Ο κύριος Σεβερίνα, εκ μέρους των σοσιαλιστών, έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η, Ουκρανία είναι μια πολύ σημαντική για εμάς χώρα, μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί περιέγραψε τέλεια την κατάσταση, αλλά και τις προσδοκίες μας επίσης. Όμως εξελέγει μια νέα κυβέρνηση με ελεύθερες δίκαιες εκλογές. Όλοι το αναγνωρίσαμε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα είναι η κατάλληλη ώρα να αφήσουμε την χώρα αυτή να δώσει τα αποτελέσματα και όχι να προδικάσουμε από τις πρώτες ημέρες και μήνε τη εκλογή τη νέα κυβέρνηση για τα επιτεύγματα ή τα μη επιτεύγματά τη. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που έχουμε εμεί εδώ πάρα πολύ γρήγορα διαιρέσαμε τη χώρα αυτή σε φιλοδυτικούς και φιλοανατολικούς. Και τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, διότι η φιλοδυτικοί δεν είναι στην εξουσία και δεν μπορούμε εμείς να αναγνωρίσουμε τη δυνατότητα των λεγόμενων φιλοανατολικών να προωθήσουν τη χώρα και να ε, εκπληρώσουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες. Σήμερα λοιπόν κύριε Πρόεδρε αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πραγματικό πρόβλημα στη συζήτηση και νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι φιλοευρωπαϊστές είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της Ουκρανίας και αυτοί οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τον ε, ευρωπαϊκού τύπου εξυγχρονισμό της χώρας. Ολοκληρώνοντας, να παρακαλέσω τους συναδέλφους να αποφασίσουν για την αναβολή του ψηφίσματος το οποίο θα εγκρίνουμε γιατί νομίζω ότι η χώρα έχει να κάνει με εκλογέ, με διαπραγματεύσει ε, και με εμά και δεν νομίζω ότι θα πρέπει εν μέσω μια πολιτική διαδικασία και πριν να έχουμε στη διάθεσή μα δεδομένα και στοιχεία για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, να συζητούμε και να αποφασίζουμε πράγματα. Πρόεδρο, ε, τώρα εκ μέρου ε, των φιλελευθέρων το λόγο έχει η κυρία Βαλάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Κύριε Πίτροπε, φαίνεται να έχουμε προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε τον ανατολικό μας γείτονα, την Ουκρανία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ουκρανία. Μια φορά συμπεριφέρεται στην Ευρώπη σαν να είναι σύμμαχος και στην άλλη φορά σαν να είναι αντίπαλος ή πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζουμε τις επιτόπιες πραγματικότητες και να βρούμε κοινά στοιχεία για να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες. Η οικονομική συνεργασία πάντα ήταν το ισχυρότερο όπλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για μεγαλύτερη ολοκλήρωση και η επιτυχία της οφείλεται από το 1956 σε αυτή την προσέγγιση. Πρέπει να συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε σε θεσμικέ και οικονομικέ μεταρρυθμίσει που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η Ουκρανία παράλληλα. Δυτή προσέγγιση. Αυτή είναι η μόνη δυνατή προσέγγιση. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν φαύλο κύκλο που θα οδηγήσει σε δημοκρατική σταθερότητα σε αυτή τη χώρα και στην Ανατολική αυτή γειτονιά. Προτεραιότητα να υποστηρίξουμε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και να επιτευχθεί μια οικονομία της αγοράς στην Ουκρανία ενθαρρύνοντας την ιδιοκτησία και μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το ΦΠΑ και προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η διαφθορά που είναι σε ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό η Συμφωνία Σύνδεσης θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο μεταρρύθμιση. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσει για να δημιουργηθεί μια πλήρη και βαθιά ζώνη ελευθέρου εμπορίου και να υποστηρίσουμε και την προσχώρηση της Ουκρανίας στην συνθήκη για την ε, ενεργειακή συνεργασία. Και η είσοδος της Ουκρανίας στον ΠΟΕ είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποδεχτεί, βήμα να αποδεχτεί η Ουκρανία τις προδιαγραφές οικονομικές της Ευρώπης. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτό το φαύλο κύκλο αμοιβέ εμπιστοσύνη και που θα είναι κάτι υποφελέ για όλη την περιοχή και για την ε, Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Βαλάν. Εκ μέρου των Πρασίνων τώρα έχει το λόγο για τρία λεπτά η κυρία Χάν για να μα παρουσιάσει τη θέση τη ομάδα τη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τις ανησυχίες για μία όξυνση και ε, για μη δημοκρατικές διαδικασίες στην Ουκρανία τις ημερίζομαι διότι Υπάρχει όλο και περισσότερο θόρυβος σχετικά με απειλές μεμονωμένων, με καταπιέσεις ε, δεσμευμένων μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων ατόμων που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, για τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών και όλα αυτά μας ανησυχούν. Αλλά ε, όσον αφορά την ελευθερία ελευθερία του τύπου ο δεν νομίζω ότι η καταπίεση ξεκίνησε με τις τελευταίες εκλογές. Σας είπα ότι όλοι οι ηγέτες στην ε, ουκρανική τη σκηνή ε, χρησιμοποίησαν την ε, αρχή για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και γι' αυτό πρέπει όντως να ανησυχούμε. Νομίζω ότι δεν διευκολύνουμε τη θέση μας εάν ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα χωρίς ε, να αναρωτηθούμε ε, σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις στην Ουκρανία διότι διαπιστώνω ότι η επιρροή της Ρωσίας στην Ουκρανική βιομηχανία, στον τομέα της ενεργείας αλλά και σε άλλους τομείς συστηματικά διευρύνεται. Γι' αυτό και θα σας, ε, θα σας πρότεινα να μην ψηφίσουμε αύριο αλλά πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία αφού γυρίσει η αποστολή από την Ουκρανία που θα πάει την παραπάνω εβδομάδα αφού συγκεντρώσουμε στοιχεία και αφού συνανοηθούμε σε όλους τους τομείς για να δούμε ε, τι θέλει να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτή την κατάσταση. Έχω ακολουθήσει αυτή την οδό ε, ε, με φίλους από την Ουκρανία Ουκρανία από παλιά μέχρι σήμερα. Η Ουκρανία κάποια στιγμή ήταν σε πολύ καλό δρόμο. Στις ε, τελευταίες εκλογές πιστεύω ότι η διεξαγωγή ήταν δημοκρατική. Εάν όμως τώρα η κατάσταση δεν βελτιώνεται και επιδεινώνεται πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς πώς θέλουμε και αν θέλουμε να επέμβουμε και σας προτείνω πριν από την επόμενη επίσκεψη στην Ουκρανία να έχουμε αποφασίσει τη στάση μας. Νομίζω ότι θα ακουστούμε περισσότερο εάν ε, επί που θέσουμε τα ερωτήματα τα οποία συζητιούνται στο ψήφισμα και όπως σας είπα ανησυχώ έχω πολλές, ε, ε, πολλά νέα και πληροφορίες ότι η κατάσταση επιδεινώνεται αλλά δεν νομίζω ότι αν λάβουμε μία απόφαση στο πόδι και στα γρήγορα θα διευκολύνουμε την κατάσταση Σας ευχαριστώ πολύ Μέχρι των μεταρρυθμιστών ο κύριος Καμίνης και έχει το λόγο για ένα λεπτό εμείς συμμετείχαμε στην Πορτοκαλή Επανάσταση. Ήμασταν οι Ουκρανοί δημοκράτες δύσκολες, σε δύσκολες εποχές. Και στην Ουκρανία λέγαμε ότι αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε δεν συνδεόταν με συγκεκριμένη πολιτική ομάδα αλλά ήμασταν υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Να μην λησμονούμε σήμερα. ότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλω να μεροληπτούμε, θέλουμε να υπερασπιστούμε κάτι σημαντικό. Να είμαστε φερέφωνο εκείνων που θέλουν την ανεξαρτησία, δηλαδή υπέρ του ουκρανικού λαού. Και να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες στην Ουκρανία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το ψήφισμα όσο έχει δεν θα βοηθήσει τους φίλους μας στην Ουκρανία. Αυτό το ψήφισμα θα σπρώξει την Ουκρανία προς τη Ρωσία δίνοντας επιχειρήματα σε εκείνους που λέγουν ότι δεν υπάρχει θέση για την Ουκρανία στη Δύση. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία, να πιέσουμε την Ουκρανία τόσο ώστε αυτά τα πρότυπα, αυτές τις προδιαγραφές να εφαρμοστούν, αλλά να μην αφήσουμε την Ουκρανία να απομακρυνθεί και να κινηθεί προς Ανατολάς. Εκτιμώ τα όσα συνέταξε ο συντάκτης του ψηφίσματος που πολεμά για, τα, για την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όμως τα λόγια για να βοηθήσουμε την Ουκρανία. ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από την αρχή αυτής της εβδομάδος και δυστυχώς... Ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο είδα δυσάρεστες επικεφαλίδες στις εφημερίδες διότι βλέπουμε ότι στα ανατολικά της ε, Ευρώπης οι γείτονές μας φοβούνται ε, την ε, ανομία στην Ουκρανία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες τις οποίες συμπράττουν και οι πολιτικοί. Εν τω μεταξύ τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι οι μεγαλύτεροι άμεσοι επενδυτές στην Ουκρανία. Κύριε Επίτροπε Φίλε, αναγνωρίζετε την, το μέγεθος των επενδύσεων της Ευρώπης στην Ουκρανία και τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να προασπίσετε τα ε, συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων στην ε, χώρα αυτή. Θέλουμε με να προωθήσουμε την προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την οικονομική και ε, την ε, πολιτική πτυχή. Ολοκληρώντας θα δώσω το λόγο στον κύριο... Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γιαννούκοφιτς ε, πήρε την αρχή και έκτοτε ε, χάθηκαν τα δημοκρατικά επιτεύγματα. Οπότε, ε, αν αξιολογούμε την κατάσταση, βλέπουμε ότι η δημοκρατία, σύμφωνα με τις δικές μας ιδέες, δεν ισχύει επί ίδιου επίπεδου και δεν μπορεί να μεταφερθεί με τον ίδιο τρόπο σε πρώην κομμουνιστικές χώρες. Έχει μεν ε, ενισχυθεί η δύναμη του Προέδρου και έχει αποδυναμωθεί το Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, δεν υπάρχει ένα ιδεώδες σύστημα ε, υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία του τύπου και ο κύριος Γιαννούκοβιτς δεν είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί δημοκρατικά μέτρα και σταθμά υπάρχουν μένες μεταρρυθμίσεις οικονομικές για να υπάρξει ανάπτυξη στην χώρα και ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίσει. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Σέφλιν. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία σαφώς δείχνουν αυτό που αναφέρεται, ότι η εξουσία διαφθείρει απόλυτη, εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η ελίτ που κυβερνά ασκούσε την εξουσία από την εκλογή του Προέδρου Γιονίκοβιτς και τα περισσότερα από αυτά που έγιναν οδηγούν προς την κατεύθυνση υποστήριξης της συγκέντρωσης των εξουσιών. Και αυτό είναι πιο εντυπωσιακό αν θυμηθούμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που δώσαν Νούκοβιτ μια μικρή πλειοψηφία και έδειξαν ότι είχε ισχυρή υποστήριξη στα νότια και ανατολικά τη χώρα και μόνο. Όμω, και εδώ αυτό μα εκπλήσει όσον αφορά την πολιτική στην Ουκρανία. Τώρα υπήρχε σαφή μετακίνηση προς τον εξυγχρονισμό εναλλακτικών κέντρων εξουσίας. Τα μέσα ενημέρωσης, αντιπολίτευση, αυτονομία της κρατικής δίκησης όλα έχουν πληγεί. Κυρίως ανησυχητική είναι η μυστική αστυνομία που απέξε τη δυνατότητα να μπορεί να παρεμβαίνει εκτατικότατα στα θέματα της χώρας. Όλα αυτά είναι κακή για το μέλλον, κυρίως αν οι Ουκρανοί πραγματικά θέλουν να έχουν ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Διότι το σύστημα που δημιουργεί ο Γιαννούκοβιτς οδηγεί μακριά από την Ευρώπη και όχι προς την Ευρώπη. Το πολύ μπορούμε να πούμε για την αλλαγή είναι ότι επέφερε ένα βαθμό σταθερότητα στη χώρα, αλλά όλο και περισσότερο αυτή η σταθερότητα ε, οδηγεί σε αποτελμάτωση και κινησία. Αυτό θα φρεβιφέρει. Ο, ο Γιαννούκοβιτ σίγουρα βελτίωσε τι σχέσει εντωμεταξύ με τη Ρωσία και δέχτηκε ένα βαθμό όμως υποτέλειας στη Ρωσία και αυτό είναι κάτι καινούριο. Τώρα αν η Ουκρανική κοινωνία θα δεχτεί αυτή τη μεταμόρφωση μακροπρόθεσμα είναι θέμα ανοιχτό. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Μάρι έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε τελικά να θέσουμε το εξή ερώτημα. Τι έγινε, πραξικόπημα, στρατιωτική παρέμβαση, τι ήταν αυτό που συνέβη στην Ουκρανία. Γράφονται το βράδυ ε, κάποιες προτάσεις ε, και την άλλη μέρα λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία. Νομίζω ότι με το ψήφισμα ε, καταδικάζουμε ε, ε, λατινοαμερικανικά και αφρικανικά καθεστώτα, αυτά βέβαια δεν μπορούν να ταυτιστούν όσα συμβαίνουν στην ε, Ουκρανία. Πράγματι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μας δυσαρεστούν, αλλά τελικά τι γλώσσα θα υιοθετήσουμε απέναντι σε αυτή τη χώρα. Το λόγο της άρνησης, Νομίζω ότι ίσως να έχουμε κάποια αρνητικά αποτελέσματα και εμείς θα πρέπει να καταδεικνύουμε τα λάθη, όχι όμως τώρα και όχι με αυτόν τον τρόπο. Η Τιμοσέγκο ε, έχασε τις ε, εκλογές, είχε κάτι αλλά τις έχασε τις εκλογές σας. Ε, αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να δούμε τι κάνουν οι αρχές τώρα στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κόβαλ για 1,5 λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Φίλε για την προσέγγιση του, η οποία είναι επικοδομητική. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Ρεμπέκα Χάρνσε που μίλησε πολύ συνετά για την Ουκρανία. Όλα τα στοιχεία του ΑΣΕ δείχνουν ότι η Ουκρανία είναι η μόνη χώρα της πρώην σοβιετικής Ένωσης που μέχρι τώρα διοργάνωσε φυσιολογικές εκλογές, κανονικές εκλογές. Αυτό είναι πρόοδο. δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και πριν δε τις προσεχείς εκλογές. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ακολουθήσει το δρόμο ε, του ΕΛΚ που ουσιαστικά αντιτίθεται σε μια χώρα που έχει διοργανώσει παρόλα αυτά κανονικές εκλογές λίγο πολύ. Τώρα θέλω να στραφώ στους ε, προσκεκλημένου μα από την Ουκρανία. Η θέση τη Ουκρανίας είναι εδώ, εδώ σε αυτό το χώρο, σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό ακριβώ και εφαρμόζουμε για την Ουκρανία τα ίδια κριτήρια με τα κριτήρια που εφαρμόζουμε και στα κράτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά κράτη. Κάθε πρόβλημα, όσο μικρό και αν είναι, με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, πάντοτε θα το σχολιάζουμε εδώ. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό αδελφοί μου από την Ουκρανία. Είστε Ευρωπαίοι και πρέπει να είστε στο ύψος των ευρωπαϊκών αρχών. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω σε εσά αυτήν την έκκληση. Έχετε κάποιες αντιπαραθέσεις εσωτερικές στη χώρα σας, εμείς τις παρακολουθούμε, εσείς όμως πρέπει να είστε ενωμένοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είστε ενωμένοι απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είτε είστε πορτοκαλί, είτε είστε γαλάζιοι, είτε είστε κίτρινοι, η θέση σας είναι εδώ. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι τόσο ταχεία η διαδικασία. Εμείς όμως σα στείλουμε χείρα φιλίας. Το ψήφισμα ουσιαστικά αυτό ε, προβλέπεται για μετά τις εκλογές, αν θέλετε ουσιαστικά. Δηλαδή προβλέπουμε μια κοινή θέση. Όταν λέω κοινή εννοώ για τις δύο πλευρές, ώστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει Περάσατε δυστυχώ ε, το χρόνο αγόρης που είχατε στη διάθεσή σα, ε, Κυρία Βάιντερη. Ευχαριστώ πολύ. Η Ουκρανία είναι πολύ σημαντική αποστατική σκοπιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι για τα τεκτενόμενα εκεί. Την 1η Οκτωβρίου δεκάδε χιλιάδε Ουκρανοί διαμαρτυρήθηκαν, διαδήλωσαν στου δρόμου τη Ουκρανία κατά των μεταρρυθμίσεων των συνταγματικών που ξεκίνησε ο Γιαννούκοβιτς. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν πέρασαν μέσα από καμία δημοκρατική διαδικασία και δεν εναρμονίστηκαν με την Επιτροπή Μπένες. Και αυτό απειλεί την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί φίλοι μας ανησυχούν. Ανησυχούν για τις εκλογές και επίσης επειδή για πολιτικούς λόγους τα κυβερνώντα κόμματα χρησιμοποιούν το δικαστικό σύστημα για δικούς τους σκοπούς. Γι' αυτό το ψήφισμά μας είναι απόλυτα αναγκαίο τώρα. Η συμμαχία που κυβερνά ε, απέρριψε την πρόταση των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, ούτως ώστε η Ουκρανία να γίνει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να τεθεί αυτός προτεραιότης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει. Να βοηθήσει να επικρατήσει ελευθερία στα μέσα ενημέρωση στην Ουκρανία. Όταν ένας μεγιστάνας των μέσων ενημέρωση είναι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μιας δημοκρατικής χώρα. Πέραν αυτού, θα πρέπει να κάνουμε και κάποια θετικά βήματα. Να εισαγάγουμε εξαιρέσει από ανάγκε θεώρηση διαβατηρίων και να βοηθήσουμε στον ενεργειακό τομέα, να συνεργαστούμε εκεί, να υποστηρίξουμε δημοκρατικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυτό θα ήταν και καθήκον και περιεχόμενο του επόμενου ψηφίσματο μετά τι εκλογέ, όπου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε άλλα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία. Σα ευχαριστώ κύριε Βάιντερ. Έχω δύο συναδέλφου που θέλουν να σα απευθύνουν ένα ερώτημα, αν επιθυμείτε βέβαια να απαντήσετε. Επιθυμείτε. Κυρία Βάιντερε, επαναλαμβάνω, δύο συνάδελφοι ζήτησαν ε, την άδεια να σας υποβάλουν ε, ερώτηση. Εσείς θέλετε, επιθυμείτε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σίβιτς. Ένα απλό ερώτημα έχω. Είπατε ότι η παρούσα κυβέρνηση Ουκρανίας απέρριψε την μελλοντική προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση του Προέδρου, από ό,τι γνωρίζω, και η επίσημη επίσης δήλωση του Κοινοβουλίου για τη μακροχρόθεσμη πολιτική είναι ότι θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Ουκρανία. Δεν ξέρω, σας παρεξήγησα ή παρεξηγήσατε, σας παρεξήγησα εγώ ή παρεξήγησατε εσείς αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Κυρία Βάιντερ, μπορείτε να απαντήσετε. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Μάλιστα, θα ήθελα να τα πω πιο ξεκάθαρα τα πράγματα ίσως να μην έγινε αντιληπτή. Είπε ο Πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι πολιτική προτεραιότητα σύμφωνα με την απόφαση του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Madam Harms, you want to put a question? You 30 Έχετε 30 δευτερόλεπτα κυρία Χάρμς για να κάνετε τη δική σας ερώτηση. Ευχαρίστω θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο εφόσον τώρα έχουμε ένα κείμενο όπου υπάρχουν όλα τα σημεία ε, που μας ανησυχούν σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας και την καταστολή στην Ουκρανία ε, εφόσον υπάρχει τώρα το κείμενο γιατί να πάμε σε δύο εβδομάδες το κείμενο και να το συζητήσουμε. Καλύτερα δεν θα ήταν να περιμένουμε μετά την επίσκεψη και μετά να πάρουμε απόφαση. Γιατί ε, βάσει των εμπειριών της, ε, ε, των αποστολών μας πιο, ο πιο επικοδομητικός τρόπος να επηρεάσουμε είναι μετά την επίσκεψη. Θέλετε να απαντήσετε. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο μετά τη δική μας συμμετοχή στις συνομιλίες υψηλού επίπεδου στην Ουκρανία παίρνουμε αυτά τα μηνύματα από την Ουκρανία. Όσον αφορά την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής της Υπεύθυνης για τις εκλογές και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εάν εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, πιστεύω ότι οι περιφερειακές εκλογές θα είναι πολύ πιο δημοκρατικές. Βεβαίως μπορούμε να πάμε μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στην Ουκρανία με το ψήφισμά μας. Κανείς δεν θα μας εμποδίσει από το να ετοιμάσουμε ένα νέο ψήφισμα. Η κατάσταση όμως της δημοκρατίας επιδεινώνεται στη χώρα αυτή. Αυτό είναι γεγονός. Ε, Σας προτείνω να ζητήσετε το λόγο στο Catch the Eye δεν μπορούμε ε, να επιτρέψουμε 40 συνάδελφοι να σηκώνουν ε, τη γαλάζια κάρτα και να γίνεται έτσι η συζήτηση, γιατί ξέρετε υπάρχουν ε, συνάδελφοι που είναι γεγραμμένοι στο κατάλογο των νομιτών, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν και τελικά δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Αν θέλετε λοιπόν, εγγραφείτε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριο Βιγγένιν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έλεγα ότι η ποιότητα τη σημερινή συζήτηση δείχνει ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, ούτε χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι ούτε η κατάλληλη χρονική στιγμή ε, και για την έκρηση ψηφίσματο για την Ουκρανία, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Πριν από έξι μήνες σα υπενθυμίζω ότι η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση ελεύθερης ε, πτώσης, στο χείλος ε, του χάου. Πολιτική, οικονομική αστάθεια, ε, βαθιά κρίση ήταν τα χαρακτηριστικά. Τώρα η εικόνα είναι εντελώ διαφορετική. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα σε λίγου μήνε η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να επαναφέρει στη φυσιολογική κατάσταση τη χώρα σε πολιτική, οικονομική και οικονομική σταθερότητα. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτό δεν το αγνοούμε ούτε το αρνούμεθα, αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι σήμερα ε, υπάρχουν κάποια διορθωτικά μέτρα τα οποία έχουν ε, ληφθεί. Παραδείγματο χάρη για τον εκλογικό νόμο για κάποιε εκλογικέ διαδικασίε. Υπό αυτήν την έννοια θα ακουστεί εκεί η φωνή μα, αλλά θα ακουστεί όχι αν ε, αρθρώνουμε κραυγέ ε, συνεχώς, αλλά με άλλο τρόπο. Και γι' αυτό η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα πάει σε 10 μέρε στην Ουκρανία, νομίζω ότι ε, δεν θα κάνει κανένα καλό για το Κοινοβούλιο. Αντίθετα θα υπονομεύσει το ρόλο του Κοινοβουλίου εάν ε, δέκα μέρε πριν τις εκλογές ε, πάμε με ένα τέτοιο ψήφισμα, να έχουμε εγκρίνει ένα τέτοιο ψήφισμα. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θα είναι μια σαφή απόπειρα επηρεασμού των εκλογών. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να αναβάλουμε την έγκριση του ψηφίσματος να ζητήσουμε από του συναδέλφου μα από την Επιτροπή Κοινοβουλευτική Συνεργασία να ελέγξουν με του εκεί συναδέλφους, να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώ ε, έχετε υπερβεί το χρόνο σα, ε, αγαπητέ συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρο. Για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, ο κύριο Ουγγουρεάνου έχει τώρα το λόγο. Οι νέε Ουκρανικέ αρχέ είναι κατόνομα μόνο νέε και ακολουθούν αυταρχικέ ε, καταπιεστικές μεθόδους. στο νομικό πλαίσιο για τις επικείμενες τοπικές εκλογές ε, άλλαξαν οι κανόνες και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το Σύνταγμα άλλαξε επίσης. Μέσω και έχει επιστρέψει ένα de facto καθεστώς προεδρικό. Τα μέσα ενημέρωση και η κοινωνία των πολιτών υπό σταθερή πίεση. Η μυστική υπηρεσία τη Ουκρανία φαίνεται να ξαναζεί τι μέρε τη Σοβιετική Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, και είναι η ώρα λοιπόν να εκφράσουμε σαφώ τι ανησυχίε μα σε ένα, μέσω ενός ψηφίσματος. Οι Ουκρανικές αρχές θα πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι οι στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εγγυημένε μέσω φιλικών δηλώσεων και μόνο. Μια μη δημοκρατική κυβέρνηση, Ουκρανική κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως σε μια στατηγικά ευαίσθητη περιοχή όπως είναι ο Εύξηνος Πόντος. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής στο γύρο αυτό είναι ο κύριος Βόποτα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας διότι η κυβέρνηση ε, της ε, Ουκρανίας εφαρμόζει το κράτος δικαίου και η ε, αντιπολίτευση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην μεταδίδει ψευδείς πληροφορίες διότι λέγεται ε, ότι ε, υπάρχει παραπληροφόρηση η οποία διαψεύδεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους άρα ε, δεν πρέπει εμείς να εμπλακούμε σε αυτά τα παιχνίδια τα κομματικά δεν είναι κύριοι του ΕΛΚΑ αυτό το δικό μας κατοίκων. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά θα έχουμε την ε, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή η οποία ε, θα πάει στην Ουκρανία και κύριε Γκάλερ πάντοτε λέμε μετά τις εκλογές εάν τα πράγματα πήγαν καλά ή κακά και όχι εκ προημίου να καταδικάζουμε και να προδικάζουμε. Πρέπει να μείνουμε δίκαιοι και σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Γκάλερ. Κύριε Γκάλερ, έχετε σηκώσει την μπλε κάρτα. Ή τι, μήπως ε, δείξατε τα κέρατα κάποιου τάφου, δεν κατάλαβα ακριβώ. Λοιπόν, σας πρέπει να κάνετε μια ερώτηση για 30 δευτερόλεπτα. Θέλω ένα λεπτό όταν θα έχουμε τη διαδικασία catch the eye, οπότε θα έχω ένα λεπτό. Κοιτάξτε, όμως, αλλά έχουμε πάνω από τους διπλάσιους ομιλητές σε σχέση με που επιτρέπονται από τους κανόνες στη διαδικασία Catch the Eye, προσέλκυση της προσοχής του Προέδρου. Κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Είδατε, κάποιο ε, τελικά γράφεται και ζητά την προσοχή του Πρόεδρου και δεν είναι εδώ. Λοιπόν, κυρία Λουκασιέσκα τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάποιο που δεν γνώρισε το σοσιαλιστικό σύστημα θα καταλάβει ποτέ το, τους λαούς που γνώρισαν ένα τέτοιο καθεστώς, περιορισμό των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης και των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν θα καταλάβουν τι δρόμο έχουν ακολουθήσει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σήμερα. Δημιουργούνται ερωτηματικά. Πρέπει να λάβουμε όμω και τι μικρέ αλλά σημαντικέ αλλαγέ που έλαβαν χώρα. Όπω οι πρόσφατε δημοκρατικέ εκλογέ. Και εμεί ήμασταν μάρτυρε ω εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να καταλάβουμε τι εκατοντάδε χιλιάδε νέου Ουκρανού που βασίζονται σε εμά, στη βοήθειά μα, για να οικοδομήσουν την δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών. Είναι εύκολο να επικρίνει κανείς. Εγώ όμως είμαι Πολωνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ψήφισμα τόσο σύντομα και ιδιαίτερα πρώτων εκλογών, πρώτης επίσκεψης ε, και πολύ περισσότερον πρώτης παρουσίας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην ουκρανία. η κυβέρνηση αυτή έχει πρόσφατα εκλεγεί είναι γεγονό ότι υπάρχουν προβλήματα οφείλουμε όμω να αναγνωρίσουμε ότι εκλέγει και με δημοκρατικές διαδικασίε και να τη δώσουμε το δικαίωμα να συνεχίσει την προσπάθειά της. οποιοδήποτε ψήφισμα θα έχει έννοια εάν γίνει μετά τι αναμενόμενε εκλογέ στην ουκρανία. ευχαριστώ. Gracias. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαυρονικόλα. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Οβίρ. Μικρο, μικρο. okay, excuse me. Ε, Καλώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα ένα ερώτημα που ήθελα να απευθύνω στον καλό συνάδελφο, στην κυρία Βάιντερε μάλλον, τη συνάδελφό μου. Αλλά θα ήθελα να πω, να εκφράσω τι με ανησυχεί και τι με αγχώνει. Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα για την Ουκρανία σήμερα ή αύριο. Δεν είναι καλή, καλός χρονικός συντονισμός αυτός. Οι Ουκρανοί δεν θα μας καταλάβουν. Αυτό που έχουμε σαν σχέδιο κειμένου μπροστά μας έχει έναν τόνο που δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Δεν είναι το σωστό ύφο, δεν είναι το σωστό ψήφισμα. Και περιέχει και κάποια πραγματικά σφάλματα. Η κυρία Βάιντερ αναφέρθηκε στι επικρίσει του Προέδρου τη της Επιτροπή Βένε όσον αφορά τι συνταγματικέ τροποποίησει. Έχω μία επιστολή. Έλαβα μία επιστολή όπου εκφράζονται διάφορες ανησυχίες, την, την πίκρα, εκφράζεται πίκρα για τη συμπεριλήφθη ένα τέτοιο σημείο στο ψήφισμά μας. E, Σας ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ πως ο κύριος Βιγκάνιν ότι είναι άσχημα τα πράγματα. Είναι πολύ καλή συζήτηση. Είναι σπάνια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Και η παρέμβαση της κυρία Λουκατσεύσκα καταδεικνύει ότι ε, υπάρχουν και άλλοι σε αυτή την άποψη. Ευχαριστώ τους σοσιαλιστές, ευχαριστώ τον κύριο Σβόμποντα τον κύριο Σεβερίν και τον κύριο Μαρεξκίεβιτς, διότι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση που στη χώρα. Πριν από τις εκλογές δεν, δεν έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις άσχημες για τους φίλους μας. Ο Επίτροπος Φούλερ και η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς έχουν και αυτοί δίκιο όταν λένε ότι βλέπουμε πράγματα που μας ανησυχούν και θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα τέτοιο από την αίθουσα. Αν θέλουμε να είναι τέρι μας οι Ουκρανοί και να έρθουν να παρίστανται σε αυτή την αίθουσα που είναι επιθυμία μας για να γίνει αυτό τότε και εδώ διακόπτεται ο μιλητής. Πρόεδρε, εντός μίας εβδομάδας δεν είναι δυνατόν ε, να αλλάξετε ούτε την νομοθεσία ούτε την ε, Επιτροπή Εκλογών. Λοιπόν, ε, ε, δεν είναι δυνατόν ε, να βλέπει κανείς επειδή δεν θα κερδίσουν οι σύμμαχοί σας ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε τη δημοκρατική τάξη της χώρας. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ισχύσουν καλύτερες συνθήκες για τη δημοκρατία στη χώρα αυτή και να στηρίξουμε την δημοκρατική κυβέρνηση γιατί ίσως η Ουκρανία δεν αρέσει σε ορισμένους και εγώ είμαι υπέρ του να ε, αναβάλουμε την ε, ψηφοφορία για αυτό το ψήφισμα. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ουκρανία είναι από τους στενότερους πιθανούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Η Ουκρανία είναι πολύ εγκύτερα όσον αφορά τα πολιτιστικά στοιχεία από ότι η Τουρκία ή η Αλβανία. Οι πορτοκαλί πολιτικές δυνάμεις κέρδισαν την περασμένη φορά. Ο Γιαννούκοβιτς ήταν επιμακρών στην αντιπολίτευση πρέπει να δεχθούμε ότι ο Γιαννούκοβιτς ίσως να θυμάται την περασμένη περίοδο όταν είχε εξωστρακιστεί από τις πορτοκαλί δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια στάση ανωτερότητας απέναντί του. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε οικονομική συνεργασία μέσω οικοδόμησης ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στην κυβέρνηση ότι η αντιπολίτευση έχει θεμητή θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και θα πρέπει να εξηγήσουμε στην αντιπολίτευση ότι εάν δεν κερδίσει εκλογές διακόπτεται εδώ ο μιλητής. Κύριε Γκάλερ, ζητήσατε διαδικαστικό επειδή μου απευθύνθηκαν προσωπικά ήθελα με τη διαδικασία Catch the Eye να μπορέσω να απαντήσω για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Ομπερμάγερ. Εσείς, ε, υποπρόεδρος, δεν ε, μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε, με την δημιουργία μίας ενεργειακής ε, κοινότητος ε, έχει δημιουργηθεί μία κοινότητα η οποία με τη συμπερίληψη της Ουκρανίας θα μπορέσει να επεκταθεί ε, ανατολικά και αυτό είναι καλό. Τα τελευταία χρόνια είχαμε προβλήματα λόγω των, της διαμάχης της Ρωσίας με την Ουκρανία σχετικά με το φυσικό αέριο με τις συζητήσεις τιμών της Ρωσίας είχαμε προβλήματα και ε, στη χώρα μου την Αυστρία είχαμε μία μείωση 23% της παροχής και ακόμη και η Γαλλία και άλλες χώρες είχαν σημαντικές ε, μειώσεις της παροχής. Πρέπει όμως εδώ να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, ασφαλή παροχή ενεργείας στην Ευρώπη και να να μην ε, είμαστε ένα ανδρίκελο στο παιχνίδι των τιμών της ε, Ρωσίας ε, και να εξασφαλίσουμε την τροφοδότηση των κρατών μας. Η κυρία Βέλτσεβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υποστήριζε την Ουκρανία στο δρόμο που ακολουθούσε προς τη δημοκρατία και στην εφαρμογή του κράτους δικαίου και σαν μια χώρα που μοιράζεται κοινέ αξίε μαζί μα. Σε οποιαδήποτε δημοκρατία οι εκλογέ είναι ένα είδο θερμόμετρο. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τη σταθερότητα των θεσμών, τη δημοκρατική διαδικασία, την οριμότητα των πολιτικών κομμάτων και τη κοινή γνώμη. Καλωσορίζουμε την ιδέα σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να καλέσει παρατηρητές για τις εκλογές, η συμμετοχή τους σίγουρα θα συμβάλλει στην ε, επικράτηση δημοκρατίας στις εκλογές και σε καλύτερη ουδετερότητα όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών στην Ουκρανία. Θα πρέπει η Ουκρανία να εγγυηθεί την ισορροπία των δυνάμεων. Η Ουκρανία μπορεί να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις της. Η κοινή γνώμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα εγγυηθούν τη μελλοντική επιτυχία. Κυρία Χιούτε. Ευχαριστώ πολύ. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα ο Ουκρανός Πρόεδρος ήρθε στη χώρα μου, τη Λιθουανία, για επίσκεψη και για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε ότι στόχος της Ουκρανίας είναι η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμφίβολα για να γίνει αυτό θα περάσουν πολλά χρόνια. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες, ε, πολλή δουλειά, μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς, στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς ή της καταπολέμησης της φτώχειας. Συμφωνώ όμως με τους συναδέλφους που είπαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εμείς δεν θα πρέπει εδώ να ψέξουμε την Ουκρανία ούτε να της κλείσουμε την πόρτα διότι έχει θέση εδώ στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πρέπει λοιπόν να συνομιλούμε με την Ουκρανία ως εταίρο και επίση όρις. Κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ουκρανία είναι μια μεγάλη, μια σημαντική χώρα, εταίρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σίγουρα έχει ένα ευρωπαϊκό μέλλον και θα ήταν αντιπαραγωγικό μια χώρα με τέτοια περίπλοκη εσωτερική δομή και δύσκολη ιστορία να αναφέρεται σαν αντικείμενο ιδεολογικών διαμαχών και σταθμίσεως υπέρ και κατά στις συζητήσεις μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε ισορροπημένη και προσεκτική προσέγγιση και όπως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου διενεργούνται δημοκρατικές εκλογές είναι δυσαρεστημένη η αντιπολίτευση άμα χάσει την εξουσία. Θα της δοθεί όμως μια άλλη δυνατότητα στο μέλλον σε μελλοντικές εκλογές. Γι' αυτό δεν είναι καλό να ακούμε μόνο στα επιχειρήματα της μίας πλευράς και θα πρέπει να εμπιστευτούμε την σοφία τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός δημοκρατικός εταίρος μας και προσλέπει στη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αλλά πιστεύω ότι ε, θα πρέπει το ψήφισμα αυτό να μην υποβληθεί πριν από τις εκλογές και η ομάδα μου έχει κάνει ορισμένες τροπολογίες διότι υπάρχει η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς λόγους οι δυνάμεις ασφαλείας. Παρακολουθούμε όμως προσεκτικά τη διαδικασία αυτή. Ο κύριος Γιαννούκοβιτς, ο πρόεδρος τώρα πιέζεται και υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών στη χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή. Έχω ακουδεί τους αριθμούς αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να επέμβουμε στις εσωτερικές εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας γιατί αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το Κοινοβούλιο. Η κυρία Κολάς Χαλοβίνσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ίδια επιχειρήματα είχαν αναφερθεί και πριν τις προεδρικές εκλογές όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διερωτώμεθα για το κατά πόσο θα σκόπιμο ένα ψήφισμα και ποια θα ήταν η θέση μας έναντι των δεκτενομένων στην Ουκρανία πριν τι εκλογέ Αποφασίσαμε να συντάξουμε ένα ψήφισμα μετά τι εκλογέ. και αυτό έγινε. Καλούμε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης. Κάποιοι μήνες πέρασαν έκτοτε και βλέπουμε σήμερα ότι τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Λοιπόν, αυτό που είναι το σημαντικότερο για να παγιωθεί η δημοκρατία στη χώρα αυτή είναι να γίνουν σωστά οι τοπικές εκλογές. Να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα. Και γι' αυτό είμαι υπέρ του ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τη ε, διαδικασία προσέλκυση της προσοχή του Προέδρου θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει μετά τις ε, παρεμβάσει των διαφόρων συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τρία μέρη θα έχει παρέμβασή μου. Πρώτα απ' όλα, θα απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα του συναδέλφου Μπέλντερ για τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα στην Ουκρανία. Αυτό είναι σαφές για τον τομέα αυτό. Έχω αρκετές φορές ε, λάβει το, ε, δεχθεί το ίδιο ερώτημα είτε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεση, είτε σε διάφορε άλλε συναντήσει. Και την τελευταία φορά ετέθη το ζήτημα και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως είναι ο νόμος για τις προμήθειες. και τη δυνατότητα ενδεχομένως τροποποίησης αυτού του νόμου, κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση επί του παρόντος στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου επίσης πρέπει να γίνουν περισσότερα. Με πολύ ενδιαφέρον βέβαια έχουμε παρακολουθήσει και την ε, περίπτωση της ε, Μίταλ. Τις τελευταίες ημέρες περισσότερα πρέπει να γίνουν και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τα ζητήματα ΦΠΑ που και αυτό είναι ένα καρθόδες ζήτημα ε, για τις επιχειρήσεις μας. Με τις επαφές που έχουμε τις Ουκρανικές αρχές, ε, τις τακτικές επαφές που έχουμε με επιχειρηματίες από την Ουκρανία, στόχος μας είναι να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων επενδυτών και επιχειρηματιών. Δεύτερον, Η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Η διαδικασία αυτή που έχουμε ξεκινήσει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας αφορά το ευρωπαϊκό ουσιαστικά μέλλον της Ουκρανίας. Είναι κάτι που είναι χρήσιμο και αποφελές ορισμένες φορές Αλλά αν θέλουμε στην Ουκρανία να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάσταση, χρειάζεται η χώρα αυτή τη βοήθειά μας. Και κάποιες φορές πρέπει να ελέγχουμε το τι γίνεται εκεί και αυτό που άλλωστε αναμένουν από εμάς. Αυτό το οποίο όμως δεν χρειάζεται είναι να παρασυρθούμε σε μια σφαλμένη συζήτηση. Σταθερότητα ή προσήλωση σε κάποιες αρχές και αξίες για παράδειγμα. Και έρχομαι στην τρίτη δέσμη ζητημάτων. Ποιος είμαι εγώ που θα μπορούσα να σχολιάσω το σχέδιο ψηφίσματος με το Κοινοβουλίου. Παρόλα αυτά, το γεγονό ότι η συζήτηση αυτή συνέβη, νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι ένα πολύτιμο μήνυμα που εκπέμπουμε. Οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου θα μεταβούν σύντομα στην Ουκρανία και τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα θα τα μεταδώσουν στους εκεί ανθρώπους. Και αυτό είναι σημαντικό μήνυμα. Όπως και αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ε, μήνυμα. Περιμένουμε όμως και από τους Ουκρανούς μηνύματα. Και ένα από αυτά θα, δοθούν, θα δοθεί την 31η Οκτωβρίου στις εκλογές. Θα δούμε αν θα επανεπιβεβαιωθεί η δημοκρατική πορεία της χώρας. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Όπως προβλέπει το άρθρο 151.1 για επί προσωπικού θα έχει το λόγο ο κύριος Γκάλερ. Θα τον παρακαλέσω όμως ε, να είναι πάρα πολύ σύντομος και να περιοριστεί στο προσωπικό αυτό ζήτημα το οποίο τον αφορά. Ευχαριστώ. Ε, ήθελα να αντιδράσω στα αυτά που είπε ο κύριος Σουόμποντα γιατί είπε κάτι που δεν ήταν σωστό διότι εμείς στο ψήφισμά μας είχαμε αναφερθεί σε, σε μια λανθασμένη αναφορά στην Επιτροπή της Βενετίας γι' αυτό και δεν περιελήφθη πλέον στο ψήφισμα άρα δεν είναι αντικείμενο της συζητήσεως. Θα ήθελα όμως να μας πείτε σαφώς σαν σοσιαλιστική ομάδα διότι αναφερθήκατε γενικά στο κράτος δικαίου αλλά δεν ε, είπατε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν επιτρέπεται ε, να συμμετάσχουν στις εκλογές διότι εφόσον ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο μπορούμε να το κατακρίνουμε και πριν τις εκλογές διότι δεν καλύπτει τις ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μπορεί πάντοτε δυνάμει το ίδιο άρθρο 151.1 ο κύριος Φόποντα να απαντήσει. Παρακαλώ να μείνετε κι εσείς ε, επί προσωπικού, να μην ε, επεκταθείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να γίνει τώρα μία αντιπαράθεση δύο τόμων, αλλά εν ονόματι της πολιτικές ομάδες είπα ότι ε, υπάρχει μία, ένας έλεγχος από τις μυστικές υπηρεσίες, το είχα πει και στον Αντιπρόεδρο Αζέροφ. Πρέπει λοιπόν από κοινού σαν ευρύτερη κοινότητα να κάνουμε κάνουμε και να διατυπώσουμε ένα ψήφισμα αντί να έχουμε στενές πλειοψηφίες όπως συμβαίνει τώρα. Ευχαριστώ. Με την παρέμβαση αυτή ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη συζήτηση αυτή από τους φιλελευθέρους, από την Ενωτική Αριστερά, από τους Πρασίνους, από τους Σοσιαλιστές, από τους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές και από το ΕΛΚΑ συγκεκριμένα. Εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση του θέματος και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το μεσημέρι. Έχουμε στη διάθεσή μας 5-6 ε, λεπτά για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πιούμε λίγο νερό και στις 6 ακριβώς ε, θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο που είναι η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς αγαπητοί συνάδελφοι. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien.